να υπάρχει κάτι το απτό και να μπορέσουν όλοι οι Ευρωπαίοι να ζουν με σωστό υγειονομικό επίπεδο. Σα ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Με αυτή την παρέμβαση ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτού του θέματο. Η ψήφιση των αντίστοιχων προτάσεων ψηφίσματο θα γίνει αύριο το μεσημέρι 12.00. Και περνάμε στην ακόλουθη έκθεση, που είναι η έκθεση της κυρίας Ζολή για τη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης ε, στα φορολογικά θέματα. Ως εισηγήτρια θα λάβει τον λόγο η κυρία Ζολή, που επιπλέον είναι και η πρόεδρός μου στην Επιτροπή Ανάπτυξης, ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή μας. Έχει τον λόγο η κυρία Ζολή, τέσσερα λεπτά. Oui, monsieur Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με κάποια ικανοποίηση σας υποβάλλω σήμερα αυτή την έκθεση για την φορολογία και την ανάπτυξη. Πραγματικά πρόκειται για ένα καθοριστικό στάδιο ενό μιας μάχης που αρχίσαμε να δίνουμε εδώ και καιρό. Και ε, σήμερα διεξαγάγεται στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου. Να ευχαριστήσω του συναδέλφου από την Επιτροπή Ανάπτυξη, με του οποίου ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική συνεργασία. Ελπίζω ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί αύριο κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορία. Ε, ε, με την ε, απειλή τη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, την αύξηση των τιμών των τροφίμων, οι αναπτυσσόμενε χώρε περισσότερο από ποτέ χρειάζονται την πραγματικές και ουσιαστικές πηγές χρηματοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο διεθνούς κρίσης, το να κινητοποιήσουμε τα φορολογικά μέσα περισσότερο από την απτυξιακή βοήθεια είναι ένα πραγματικό εργαλείο και μια πρόκληση. Διότι τα φορολογικά συστήματα που θα είναι αποτελεσματικά θα επιτρέψουν όχι μόνο να χρηματοδοτηθούν οι δημόσιε υπηρεσίε που είναι απαραίτητε, αλλά και την ε, διαφανή και υπεύθυνη χρήση των ε, δημόσιων κρατικών κονδυλίων. Αυτό θα βρίσκεται στη βάση ενός υπεύθυνου δημοκρατικού συστήματος. Έτσι θα ε, συγκεντρώνονται φόροι ισότιμοι, διαφανείς και δίκαιη, χωρί ε, να σημαίνει ότι θα καταργήσουμε κάθε είδους βοήθεια προς την ανάπτυξη. Απλώς θα πρέπει τα κράτη-μέλη να φροντίσουν να μην μειώσουν και το ποσοστό του ΑΕΠ τους που αφιερώνεται στην αναπτυξιακή βοήθεια. Σίγουρα η αναπτυξιακή βοήθεια δεν είναι τέλεια, δεν ε, σημαίνει ότι δεν επιδέχεται βελτιώσεων, όμως ε, έχει πληγεί σοβαρά από τι ανάγκε, τι καινούργιε που έχουν δημιουργηθεί με την οικονομική κρίση και τι κλιματικέ αλλαγέ. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να επαναθεωρήσουμε την πολιτική μα, ώστε να έχουμε ε, φορολογικά συστήματα αποτελεσματικά, στα οποία να συμβάλλουν και οι πολυεθνικέ επιχειρήσει ε, με του πόρου του και να επιτρέψουν στι αναπτυσσόμενε χώρε να πάρουν την σωστή κατεύθυνση προ την ανάπτυξη, να μειώσουν την φτώχεια, να εκμεταλλευτούν ε, πόρου τελωνιακού και τελικά να γίνουν αυτόνομοι ώστε να μην χρειάζονται την βοήθεια από τους άλλες χώρες. Προκειμένου να είναι αποτελεσματικά λοιπόν τα, φορολογικά τους συστήματα πρέπει να δούμε τι φόροι τους επιβάλλονται και τι επιτόκια από τους φορείς του Bretton Woods ε, και επίσης κατά πόσον επιτρέπονται ακόμη η φορολογική παράδοση. Έχουμε εδώ τεράστιες απώλειες φορολογικών εσόδων ετησίως τουλάχιστον δεκαπλάσια από το ποσό αναπτυξιακή βοήθεια που δίνεται από τι πλουσιότερε χώρε προ τι αναπτυσσόμενε. Εδώ θυμίζονται κατευθυντήρε γραμμέ του ΩΣΑ, που όμω δεν είναι καθόλου αναγκαίε και κάποιε φορέ γίνονται και επικίνδυνε. Διότι επιτρέπουν μη ε, μορφέ ε, μη, που δεν οδηγούν στην καλή συνεργασία, με γκρίζου καταλόγου, με συμφωνίε που δεν προβλέπουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και δημιουργούν μια ε, ψευδέστηση νομιμότητας επιτρέποντας φορολογικούς παραδείσους και βλάπτοντας ε, το σύστημα των κρατικών εσόδων τόσο του Βορρά όσο και του Νότου. Η εξάλληψη των φορολογικών παραδείσων είναι μια, ένα στάδιο απαραίτητο για την ανάπτυξη των χωρών αυτών και πρέπει να είναι μια πρωτοβουλία απαραίτητη ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ να αναλάβει τι ευθύνε τη. Όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε πρέπει να προβλέψουν νομοθεσία σαφή και δεσμευτική που να συνοδεύεται από πραγματικά ε, μέσα επιβολής κυρώσεων, ώστε να σταματήσει ε, η ύπαρξη των φορολογικών παραδείσων να γίνεται ένα μέσο μαζική καταστροφή των ε, αναπτυσσόμενων φτωχότερων χωρών. Θα πρέπει εδώ η εκμετάλλευση των ε, εσόδων και η μεταφορά τεράστιων ποσών να σταματήσει να είναι κλασική πρακτική ακόμα και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που ε, εποφελούνται από την ύπαρξη αυτού του συστήματο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα διαφανέ και σαφέ που να μην ε, ε, επιτρέπει στι επιχειρήσει, είτε είναι πολυεθνικέ είτε διακρατικέ, να μην δηλώνουν τα πραγματικά του έσοδα, αλλά να υποχρεούνται να το κάνουν αυτό και να μην μπορούν να μεταφέρουν τα έσοδά του σε άλλε βάσει πολύ σημαντικό, ένα ε, απαραίτητο βήμα για την ε, καλύτερη ε, διαβίωση των πληθυσμών του Νότιου Ημισφαιρίου και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξαπιστία ευχαριστούμε κυρία Ζαλή. Ευχαριστούμε κυρία Ζαλή. Έχουμε πέντε ή τέσσερι συναδέλφου που θέλουν να παρέμβουν. Πρώτα απ' όλα η κυρία θελουν να παρεμουν Ένα λεπτό γνωρίζετε καθένα. Θα αφαιρώ τον λόγο όταν θα ξεπερνάτε το όριο. Κυρία Βατσέσκου, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μέσα στην τωρινή οικονομική κρίση η χρηστή διακυβέρνηση είναι κάτι απαραίτητο και μέσα και έξω από την Ένωση. Θα έπρεπε να σας πω ότι κάθε χώρα έχει την ευθύνη να αποφασίζει μόνη της τη φορολογική της πολιτική και επομένως δεν πρέπει να επιβάλλουμε ούτε φραγμούς ούτε τίποτε άλλο παρά μόνο συνεργασία. Η καταπολέμηση το, της φοροδιαφυγής και των παραδείσων είναι επίσης κάτι το απαραίτητο γιατί ενθαρρύνει το οικονομικά εγκλήματα και οδηγεί σε άδικη κατανομή των φορολογικών εσόδων. Άλλο μέτρο θα ήταν η καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών μελών. Επίση, απαραίτητο είναι να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των αναπτυσσομένων χωρών στα αρμόδια διεθνή. Σα ευχαριστούμε, κυρία Βασέσκου. Η κυρία Βέσλοντ, παρακαλώ, έχει τον λόγο. Eh, Όχι. Αποσύρεται. Τότε θα λάβει τον λόγο η αγαπητή κυρία Κέλλερ, παρακαλώ. Η φορολογία είναι πολύ σημαντικό ζήτημα όταν μιλάμε για αναπτυξιακή πολιτική. Είναι σημαντικό για την πολιτική μας συνοχή προκειμένου να έχουμε ανάπτυξη χωρί φορολογικά εισοδήματα και διαφάνεια προ του φορολογουμένου, δεν θα είμαστε ποτέ συνεπεί ε, προ του αναπτυξιακού μα στόχου σε μια τόσο δύσκολη στιγμή. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την έκθεση αυτή και ελπίζουμε ότι δεν θα αποδυναμώσουν ε, του στόχου τη έκθεση αυτή στα κάτι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εδώ πρέπει να εντοπίσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν πολλέ ελλείψει, όπω οι κατευθυντήριε γραμμέ του ΩΣΑ, που δεν ασχολούνται με τον αντίκτυπο του φορολογικού ανταγωνισμού ή των φορολογικών εσόδων. Εδώ θέλουμε να υπάρχει συμμόρφωση με τι συνθήκη τη Λισαβόνα. Θέλουμε να είμαστε συνεπεί ω του πολιτικού μα στόχου. Πρέπει λοιπόν τώρα να αναλάβουμε δράση. Γι' αυτό σα στηρίζουμε να στηρίξετε την έκθεση αυτή πλήρω. Ευχαριστούμε κυρία Κέλλερ. Τελευταίο αγορητή σε αυτό το σημείο θα είναι ο κύριο Φερέιρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, ενώ είναι σημαντικό και αναγκαίο στοιχείο, δεν πρέπει να αγνοεί το γεγονός ότι η φορολογική πολιτική είναι θεμελιώδες ε, εργαλείο της πολιτικής ε, και της κοινωνικής πολιτικής με καθορισμούς ε, σαφών κριτηρίων. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαγάγει την αποκαλούμενη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα, όπως πολύ καλά λέει η συγγήτρια. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ξεχωριστή κατάσταση και οι ανάγκε των αναπτυσσόμενων Δύο παρατηρήσει σε σχέση με δύο καυτά θέματα. Πρώτον, τα οι αποκαλούμενε εταιρικέ συμφωνίε οικονομικών εταίρων. Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται στα αναπτυσσόμενα κράτη ε, με μεγάλε αντιστάσει που δείχνουν από πλευρά του, από πλευρά μα, ε, η ε, επιβολή αυτή αυτών των πολιτικών για την φορολογία. Βλέπουμε ότι οι φορολογικοί παράδεισοι εξακολουθούν να υπάρχουν με απώλεια 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τι αναψώμενες χώρε. Είναι δύο παραδείγματα που δείχνουν τι συμβαίνει εδώ σε στον τομέα αυτό για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σε ευχαριστώ κύριε Φερέρα. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση με την παρέμβαση τη κυρία Επιτρόπου, τη κυρία Δαμανάκη. Παρακαλώ Επίτροπε, αν θέλετε να παρέμβετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματο Κομισιόν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα την Επιτροπή Ανάπτυξη για την έκθεση αυτή. Με χαρά διαπιστώνω ότι η κυρία Εύα Ζολή στην έκθεσή της προσθέτει επιχειρήματα στη, σε εκείνα της ε, ανακοίνωσής μας και επίσης θέτει ορισμένους πάρα πολύ φιλόδοξους στόχους που αποτελούν πολύτιμες συμβουλές για την Ευρωπαϊκή Ένωση η κινητοποίηση εσωτερικών πόρων είναι κάτι ουσιώδες για να μειωθεί η ανέχεια να υπάρξει καλύτερη ή χρηστότερη διακυβέρνηση και να επιτευχθούν οι στόχοι της χιλιετίας. Πρέπει να βελτιωθεί η συνέργεια μεταξύ της φορολόγησης και των αναπτυξιακών μέτρων ώστε όλες οι χώρες να μπορέσουν να έχουν καλύτερη διοίκηση και καλύτερο φορολογικό σύστημα. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Εγώ προσωπικά εντυπωσιάστηκα από τους αριθμούς σας που έλεγαν ότι το ποσοστό φοροδιαφυγής είναι 10 φορές ψηλότερο από ότι η βοήθεια που χορηγείται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Πρέπει λοιπόν ταυτόχρονα να πετύχουμε δύο στόχους. Πρώτον να στηρίξουμε πιο αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικής φορολόγησης και δεύτερον να πετύχουμε μία, ένα καλύτερο διεθνές και πιο συνεργατικό φορολογικό περιβάλλον ώστε να μπορέσουν οι χώρες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφύγη και τον φορολογικό ανταγωνισμό. Αθέμητο. Η έκθεσή σας αναφέρει πολύ σωστά ποια είναι τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης του εμπορίου και δηλώνει ρητά ότι δεν αρκεί να υπάρξουν ορισμένες απαγορεύσεις. Θα ήθελα να δω ποια προβλήματα είναι τα πραγματικά που αντιμετωπίζουμε. Καταρχήν, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουν οι φορολογικές μεταβάσεις μέσω του λεγόμενου capacity building με περιφερειακές πρωτοβουλίες και καλύτερη συνεργασία και ενωσιακός και διεθνώς. Για το άλλο θέμα, ε, η Κομισιόν θεωρεί τη φοροδιαφυγή και τον αθέμητο φορολογικό ανταγωνισμό σαν τεράστιους φραγμούς για την καλύτερη κινητοποίηση των υπαρχόντων πόρων. Γι' αυτό θέλουμε να βοηθήσουμε και τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά και να προωθήσουμε καλύτερη διεθνή συνεργασία σε φορολογικά θέματα. Τελεία. Πολλά έχουν γίνει ήδη από την εποχή της πρώτης μας ανακοίνωσης. Έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα με την οικονομική σας στήριξη του Κοινοβουλίου. Αυτά που χορηγήσατε το 2010, 708 εκατομμύρια, μας βοήθησαν να προωθήσουμε μια καλύτερη φορολογική διαχείριση με δραστηριότητες όπως τεχνικά σεμινάρια, για αφρικανικές χώρες ε, στήριξη των εξορυκτικών διαδικασιών και συνεργασία με τον ΟΗΕ για την κινητοποίηση εσωτερικών πόρων. Επίσης θα χορηγήσουμε τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή συμφωνιών ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών και προετοιμάζουμε ανακοίνωση για να όπου θα αξιολογούμε κατά πόσον δεν θα μπορούσαμε χώρα με τη χώρα να υπάρξει μία υποχρεωτική αναφορά πληροφοριών κάθε χρόνο. Έχει γίνει μία πρώτη δημόσια συζήτηση και διαβούλευση και τώρα θα κάνουμε την αξιολόγηση της πράγμα το οποίο θα βοηθούσε ίσω τι αναπτυσσόμενε χώρε να καταπολεμήσουν αποτελεσματικότερα τη φοροδιαφυγή. Θέλω ειλικρινά να σα ευχαριστήσω για την στήριξή σα και είμαι πεπισμένη ότι πολύ πρόοδος μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η φορολογική διαχείριση. Χαίρομαι δε ιδιαίτερα γιατί τα θέματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και στα προγράμματα του Z20 και Z8. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Η ψήφιση επίσης και της πρότασης ψηφίσματος που έχει κατατεθεί από την Πρόεδρο Ζολή όπως είπα θα ψηφιστούν αύριο το μεσημέρι 12.00 και περνάμε